η δραστηριότητα ασύμβατη με αυτή του Ευρωβουλευτή. Πήρα επίσης από την ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τις αιτήσει για τη συμμετοχή της κυρίας Κοέβιους στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία. Έχετε παρατηρήσει όχι. Περνάμε λοιπόν τώρα